Ευχαριστώ τους πάντες. Ελπίζω ότι από μεθαύριο θα έχουμε έναν κανονισμό γύρω ε, σου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μέλτερ. Η συζήτηση για το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για την αναστολή της Συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Uh, Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μάλστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω σχετικά με τις δράσεις που αποφάσισα να, ε, ε, να, να αναλάβω μετά από τις αποκαλύψεις του τύπου σχετικά με την συμφωνία SWIFT. Στις 24 Σεπτεμβρίου Συναντήθηκα πολλούς από εσά στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και σας ενημέρωσα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο προφανώς δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Οι συζητήσεις ήταν ε, ε, πολύ χρήσιμες και βοήθησαν να διευκνιστούν διάφορα θέματα. Από τότε που ε, εμφανίστηκαν οι πρώτες σχετικές πληροφορίες στον τύπο, αμέσως ανέλαβα δράση. Όπως σας είπα και τότε, τον Ιούλιο έστειλα την πρώτη επιστολή στους ομολόγου, μου στη ΣΥΠΑ και στι 7 Σεπτεμβρίου τηλεφώνησα τον κύριο, Κοέν και του είπα ότι περιμένω ουσιαστικές πληροφορίες για τις ε, υποτιθέμενες παρακολουθήσεις. Την επόμενη μέρα του έστειλε μια επιστολή που ζήτησε ανοιχτές διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 19 της Συμφωνίας TFTP. Όπως ξέρετε αυτή είναι η διαδικασία που ρυθμίζεται μέσα στη Συμφωνία όταν υπάρχουν τέτοια ε, ζητήματα, ερωτήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Απαντώντας στην επιστολή μου, και την κοινοποίησα ε, την ε, επιστολή αυτή στην Επιτροπή Λίμπε στις 23 3 Σεπτεμβρίου, οι αρχέ των ΗΠΑ έδωσαν κάποιε εξηγήσει, αλλά κάποια σημαντικά θέματα παραμένουν αναπάντητα. Γι' αυτό σήμερα, ε, αυτή τη Δευτέρα, ε, τη Δευτέρα που μα πέρασε, ε, συναντήθηκα με τον κύριο Κοέν στι Βρυξέλλε και παρά του περιορισμού έγινε μια ανοιχτή συζήτηση και διευθυνθήκαν αρκετά σημεία. Στην συζήτηση αυτή, ο κύριο Κοέν δήλωσε ρητά ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία αυτή, οι ΗΠΑ δεν συνέλεξαν ε, οικονομικά, ε, οικονομικές πληροφορίες μέσω του SWIFT. Ε, κατά την περίοδο αυτή δεν συλλέχθηκαν τέτοιες πληροφορίες και επέμεινα να επιβεβαιωθεί και γραπτός αυτή η πληροφορία. Επίσης, συζητήσαμε με αρκετές λεπτομέρειες πιθανότητα οι να παίρνουν ε, σε κάποιο συγκεκριμένο φόρμα οικονομικές πληροφορίες μέσω του SWIFT ε, μέσω των, για, για οικονομικές συναλλαγές. Ε, και ζήτησα εξηγήσει και το κατά πόσο μια τέτοια πρακτική θα ερχόταν σε σύγκρουση με την PFTP. και Λένε οι αρχές, τον είπα, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε η συμφωνία PFTP. Κάποιες διευκρινήσεις χρειάζονται ακόμα όμως να δοθούν πριν να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας. Το να ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ είναι ε, στην ε, πρώτη προτεραιότητα της ε, ατζέντα μου. Θα γίνει η πλήρης αυτή διευκρίνηση στο άμεσο μέλλον και θα σας κρατήσω ενήμερους για το τελικό αποτέλεσμα την έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε και τώρα οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το συνάδελφο Δίας Δεμέρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προηγούμενη Ολομέλεια, στη συζήτηση για τη μελλοντική στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, είχα υπογραμμίσει ότι για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Σήμερα θέλω επίσης να υπογραμμίσω το ίδιο. Τα μέσα ενημέρωσης ε, απηχούν μια πραγματική ανησυχία των πολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο ερευνούμε και προσπαθούμε να βρούμε ε, αποδείξεις ε, κατασκοπίας η οποία θα μας ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επαρκείς αποδείξεις. Οι αρμόδιες αρχές, τόσο η κυρία Μάλστρομ όσο και ο διευθυντής της Europol έχουν δηλώσει και επανέλαβε σήμερα η κυρία Μάλστρομ ότι ότι τα γεγονότα αυτά δεν έχουν αποδειχθεί. Ε, εν ώψη αυτής της εύλογης ε, αμφιβολίας ε, δεν θα ήθελα να αναστάλει η Συμφωνία SWIFT. Το πρόγραμμα παρακολούθησης τη της τρομοκρατίας είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των τρομοκρατικών ομάδων. Η υπόθεση Breivik στην ε, Νορβηγία ε, διευκρινίστηκε και διαλευκάνθηκε πολύ γρήγορα μέσω της ε, συνεργασίας στο πλαίσιο της TFTP. Η σύμβαση άλλωστε αναφέρει ρητά το τι πρέπει να γίνει κάθε φορά που ένα μέρος παραβιάζει τη συμφωνία. Σίγουρα όμως δεν αναφέρει ότι μια απόφαση μπορεί να, για την αναστολή της ε, συμφωνίας μπορεί να ληφθεί ε, μονομερός. Θα πρέπει μέσω των τρόπων που προβλέπει η σύμβαση ε, να γίνει συζήτηση για να διορθωθούν οι αδυναμίες. Η ανησυχία που έχουμε για μια ενδεχόμενη ε, παραβίαση των δικαιωμάτων μας και της ιδιωτικής μας ζωής είναι εύλογη ε, και νόμιμη. Ε, γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε να αναζητούμε την αλήθεια, ερευνούμε χωρίς να βιαστούμε. Θα ήταν μάλλον ένας κίνδυνος δεν διορθώνεται δημιουργώντας άλλους καινούριου κινδύνους χωρίς να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχει μπλε κάρτα για σας κύριε Ντεμέρα από τον συνάδελφο Στογιάννοφ. Yes, colleague, Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ντίας Ντεμέρα. Πώς γνωρίζετε κύριε Ντεμέρα ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει παραβιαστεί. Επειδή το είπε η κυρία Επίτροπο, τι θέλετε να, πει, τι θέλετε να της πει ο κύριος Κοέν. Ασφαλώς και θα πει ότι δεν την έχουν παραβιάσει. Ο κύριο Ντεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Στογιάννοφ. Αν είχατε προσέξει αρκετά τα λόγια μου, δεν θα είχατε κάνει αυτή την ερώτηση. Εγώ δεν είπα αυτό που λέτε. Τι είπα. Είπα ότι υπάρχει μια εύλογη ε, αμφιβολία. Μα ανησυχούμε βέβαια, γι' αυτό το λόγο και ερευνούμε. Και είπα, δεν είναι δυνατόν με βάση μια υποψία να αναστείλουμε μια συμφωνία. Μπορούμε να αναστείλουμε μια συμφωνία αν έχουμε αποδεικτικά και αποδεικμένα στοιχεία. Η συνάδελφος Ζίπελ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Μάλστρον, θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπενθυμίσω ότι πριν από τις αποκαλύψεις είχαμε προβλήματα προς την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Για άλλη μια φορά θέλω να υπενθυμίσω ότι και πριν από την ισχύουσα τώρα συμφωνία είχαν το SWIFT οι Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν αξιοποιήσει δεδομένα του SWIFT, ε, του SWIFT στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο που τότε ενημερωθήκαμε μέσω των ε, ΜΜΕ. Τώρα όμως έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες ε, καταγγελίες από το Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οι οποίες ε, θέτουν αναμφιβόλο ε, πραγματικά όλη αυτή την συμφωνία. Εσείς αναφερθήκατε σε μια επιστολή προς τον κύριο Κον αλλά με εντυπωσιάζει η απάντηση ότι δηλαδή τα προγράμματα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα ε, θετικό, ε, είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και μια θετική απόρρεια του SWIFT που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εξασφαλίσει διαφορετικά. Δηλαδή μας λέει, μας λέει ότι δεν παίρνει δεδομένα από την Ευρώπη το SWIFT. Μα εάν παίρνουν στοιχεία από ένα τρίτο κράτος μέσω του SWIFT ε, προφανώς δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το, αυτή η συμφωνία. Ο κύριος Δίας Δεμέρα μας λέει ότι θα πρέπει να ε, δρούμε βεβαιασμένα. Οι συμφωνίες και τα όσα μας λένε τα ΜΜΕ όμως δεν είναι κάτι το πολύ πρόσφατο και θα ήθελα να ανατρέξω σε αυτά τα οποία πριν από αρκετό καιρό μας είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την απόσπαση δεδομένων σε η κατακράτηση δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει κρατεθεί η πρόταση που ακόμα δεν έχουμε δει. Άλλη μία πηγή επίκριση. Και τώρα μας λέτε ότι είναι βεβαιασμένο το να ζητήσουμε να παγώσει αυτή η συμφωνία. Όχι βέβαια. Εάν είχαμε αποδείξεις Ούτε θα, δεν θα πρέπει να παγώσει αυτή η συμφωνία, αλλά να ανακληθεί, να καταγγελθεί. Εγώ νομίζω ότι είναι η κατάλληλη μέθοδος, το κατάλληλο μέσο να παγώσει αυτή η συμφωνία για να αφήσουμε αρκετό χρόνο να διαρευνήσουμε, για να πιέσουμε επαρκώς τις ΗΠΑ και για να δούμε αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και αποδείξεις ότι έχει παραβιαστεί αυτή η συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε και εμείς και το όνομά μας και την υπογραφή μας να τιμήσουμε, ώστε να μην επιτρέψουμε και να μην επιτρέψουμε να ε, γίνεται κατάχρηση των δεδομένων ε, των πολιτών της Ευρώπης. Thank you, Chair. Κυρία Νετφέλτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η από το ΕΛΚ, ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, μας είπε μόλις ότι χρειάζονται δεδομένα και δεν πρέπει να λαμβάνουμε βεβαιασμένε αποφάσει. Μα συμφωνώ απολύτω. Γι' αυτό ακριβώ με εντυπωσιάζει το ότι δεν έχει γίνει καμία διερεύνηση τη υπόθεση. Ούτε ένα κράτο μέλο δεν ζήτησε από την ε, μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Europol, που θα έπρεπε να είναι αρμόδια για τη διερεύνηση αυτή αρχή, να ερευνήσει την υπόθεση. Δεν κάνει η κυβέρνηση της, ε, των κάτω χωρών, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος εξυπηρετητής Παύλα Σέρβερ της, ε, του SWIFT, έχει κάνει κάτι τέτοιο. Όλοι λένε, α, όχι, θα το αναλάβει μια ομάδα εργασία, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή, υπάλληλοι, οι οποίοι μεταξύ, πίσω από κλειστέ πόρτε ζητούν και βγαίνουν για να μα πούν ότι όλα πάνε καλά. Μα βεβαίω δεν έχουμε ε, αποδείξει, αλλά έχουμε σαφέστατε ενδείξει, εντονότατε ενδείξει. Και αυτέ δεν στηρίζονται στην, ε, στο λόγο τη τιμή του κυρίου Κοέν, ούτε σε κάποιε δηλώσει ε, του SWIFT, αλλά στην διερεύνηση. Πρέπει να πάμε στου εξυπηρετητέ του SWIFT και να ερευνήσουμε τι έχει συμβεί. Γιατί δεν το κάνουν αυτά τα κρατημέλη, γιατί δεν ζητούν από την Europol να ερευνήσει την κατάσταση, γιατί δεν επιμένουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιμένει γιατί δεν ζητάει να ερευνήσει η κυβέρνηση των κάτω χωρών επί τόπου, μέσα στον ίδιο το σερβερ, το τι έχει συμβεί. Αφού του άλλου δεν έχουμε κανένα λόγο πλέον να εμπιστευόμαστε του Αμερικανού, τι ΗΠΑ και αυτό δεν είναι μόνο λόγο των αναφορών στον τύπο. Έχουμε έγγραφα. Έγγραφα που έχει διαθέσει ο κύριο Σνόουντεν και δεν αρνήθηκαν ποτέ οι Αμερικανοί ότι ισχύουν αυτά. δεν είπαν ότι δεν είχαν μη ε, ε, ότι είχαν πρόσβαση χωρί άδεια στο SWIFT, αλλά λένε ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματο να το πράξουν ανά πάσα στιγμή. Αν λοιπόν τώρα εμεί θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή τη συμφωνία, ή μη τι άλλο, έχουμε το δικαίωμα να ερευνήσουμε, έχουμε το χρόνο να ερευνήσουμε. Και κυρία Επίτροπε, εκπρόσωπε του Συμβουλίου, ω ε, συνήθω με, με τη γνωστή άδεια καρέκλα, έχουμε μια πρώτη διεθνή συμφωνία η οποία δοκιμάστηκε υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας, μια πρώτη συμφωνία όπου ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του συγκοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι άπαξ και υπογράψαμε, επιταγή βέβαια είναι λευκό ήτανε, έχουμε βγει από το παιχνίδι. Αλλά μέσω της Επιτροπής, μέσω του Συμβουλίου θα μας ζητήσετε κάποια άλλη φορά να δώσουμε σύμφωνη γνώμη. Εδώ θα κρυθείτε. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο θα δοκιμαστεί η αξιοπιστία σας. Εάν λοιπόν δεν πάτε στον πυρήνα, στην ουσία αυτή η συμφωνία, αν η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν αντιδράσουν όσο οφείλουν, τότε πια το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει στο μέλλον σύμφωνη γνώμη σε αντίστοιχε συμφωνίε. Γιατί εδώ διακυβεύεται η ίδια δημοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριο Άλμπρεχτ, εκ μέρους των Πράσινων. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ε, πρέπει να σας πω ότι σοκάρομαι κάπως που ε, αισθάνεστε τόσο άνετα με αυτές τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση. Τον είπα, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο η συνάδελφος Τσίπελ. Ο κύριος Κόεν έγραψε ότι η κυβέρνηση ε, τον είπα χρησιμοποιεί την ε, TFTP για να, πα, για να αντλεί στοιχεία από το SWIFT που δεν αντλούν από άλλες πηγές, ε, όπως το είπαν επιλέξει. Αυτό είναι προφανές κατά τη γνώμη μου ότι προσπαθούν να αποφύγουν να λογοδοτήσουν για αυτό που πραγματικά κάνουν και για το κατά πόσον αυτό συνάδει με την συμφωνία SWIFT. Προφανώς όχι. Ε, και ε, αναφέρονται στην ε, αρμοδιότητα που τους δίνει η δικιά τους νομοθεσία να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει βάσιμος λόγος να αναστέλουμε αυτή τη συμφωνία και να ξεκινήσουμε μια πραγματική έρευνα. Επίσης, καμία κυβέρνηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμία ε, εθνική αρχή δεν ε, διερευνά αυτή, αυτούς τους ισχυρισμούς για μια πιθανή κυβερνοεπίθεση ε, εναντίον ε, των προσωπικών δεδομένων μέσω μιας ευρωπαϊκής εταιρείας. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να εργαστούμε ε, και να επωφεληθούμε από την ευκαιρία ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία και να ξαναδιαπραγματευτούμε του όρου ε, συνεργασία σε επίπεδο αστυνομία και δικαιοσύνη με τη ΣΥΠΑ και να είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, εταιρείε όπω η ΣΤΟΥΙΠ, θα ε, ακολουθούν και θα σέβονται του κανονισμού και την οδηγία που έχουμε σήμερα για την προστασία των δεδομένων και ότι ε, οι κανόνες αυτοί θα ε, εφαρμόζονται καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, συνάδελφος Κυρικό. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω το Κοινοβουλίο και την Επίτροπο. Πιστεύετε ειλικρινά ότι οι απειλέ αναστολή αυτής τόσο σημαντική συμφωνίας για την καταβλήση τη τρομοκρατίας είναι προς το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της δύση είναι η τρομοκρατία. Ε, το ε, MI5 θεωρεί ότι αυτή η διαρροή είναι δώρο προς τους τρομοκράτες και αν αναστείλουμε τη συμφωνία θα είναι ακόμα ένα δώρο εις βάρος της ασφάλειας Ευρώπης. Είναι πραγματικά αστείο αυτό. Εσείς λέτε ότι εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ όμως θέλω να εκπροσωπήσω αυτούς τους πολίτες που θέλουν να ζήσουν σε μια Ευρώπη ασφαλή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σίγουρα θα πρέπει η αρμόδια αρχή να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας και να ενισχυθούν οι κανόνες προστασίας των δεδομένων, αλλά αυτό ας γίνει μέσω της αναζήτησης πραγματικών στοιχείων και όχι με βάση υποψίες ή φήμες. Θα πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Κανένας δεν αρνείται ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των πολιτών μα. Αυτή είναι η δουλειά μα. Αλλά όχι θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή του και την ασφαλεία του. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω οποιαδήποτε κίνηση του Κοινοβουλίου να πάρει τέτοιου είδου ε, ε, μέτρα που θα είναι ανεύθυνα και θα θέσουν σε κίνδυνο τι διεθνεί μα σχέσει και την παγκόσμια ασφάλεια. Ή μήπω θα αναστείλουμε και όλε μα τι συμφωνίε κάθε φορά που μια εφημερίδα ε, ή ένα άτομο κάνει μια, ε, ένα τέτοιο ισχυρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νατφέλτ, έχει μια ερώτηση για σας, το δέχεστε, τη δέχεστε. Χωρίς μικρόφωνο. Θα δεχθείτε την ερώτηση, κύριε Νατφέλτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά ακούω ότι θέλετε να δείτε πραγματικά γεγονότα. Συμφωνείτε λοιπόν να ζητήσουμε μια επίσημη έρευνα από την μονάδα κυβερνοεκκλήματος της Europol και μάλιστα το κόμμα σας εκ μέρους της κυβέρνησης του ΕΒ δικαιούται να το πράξει αυτό εάν δεν εμπιστεύεστε εμάς, αν δεν εμπιστεύεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον εμπιστεύεστε την Europol. Και δεύτερον, λέτε ότι είναι απαραίτητο το σύστημα αυτό για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όμως ο Υπουργός Κορν μέσα στην επιστολή του αναγνωρίζει ο ίδιος ότι χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για θέματα άσχετα με τρομοκρατία. Είστε σύμφωνος με το χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ τα δεδομένα για θέματα άσχετα με την τρομοκρατία. Κύριε Κίρκοπ. Πάντα μου σηκώνει την μπλε κάρτα, Σόφη. Και μπορώ να σου πω το εξής. Νομίζω ότι η αρμόδια αρχή πάντοτε θα πρέπει να διερευνά υπενιγμού ή ισχυρισμού. Εκεί που. και δεν έχω καμιά αντίρρηση σε αυτό. Εκεί που έχω αντίρρηση είναι στη μεροληπτική αυτή προσέγγιση που βλέπω να ε, αναπτύσσεται όποτε γίνονται καταγγελίε και μάλιστα μέσω καταδίκες εκφράζονται κατά μια χώρα ή κάποιου μέρου χωρί καμιά αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων ε, ε, και αυτό συμβαίνει όλο και πιο συχνά στο κοινοβούλιο και πρέπει να πω γιατί με ενδιαφέρει το θέμα και θα ρωτώ αυτόν εμπλεκόμενο ότι είναι κάτω απαράδεκτον. Συνάδελφος Ένστε. Κυρία. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Σήμερα συνεχίζουμε τα ενηγματάκια μας για το SWIFT, τις ερωτήσεις τι θα μάθουμε, τι δεν θα μάθουμε. Τελικά δεν μαθαίνουμε όμως τίποτα, δεν, δεν κατατίθεται καμία αλήθεια στην τράπεζα, δεν ε, έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά ε, με ε, των θυρών συζητήσεις με κρυφές ε, και απόρριτες πληροφορίες. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να κοιτάξουμε να σταματήσουμε τη λειτουργία του SWIFT αφού υπάρχουν αυτές οι σοβαρές ε, ενδείξεις ε, και ισχυρισμοί μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τις ΗΠΑ. Και από την άλλη μας λέτε ότι δεν χρειάζεται γιατί έχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει συμβεί κάτι κακό. Η επιστολή είναι το αποδεικτικό σας το στοιχείο, πάνω σε αυτό στηρίζεστε. Τι είδους έρευνα έχετε κάνει, τι είδους αποδείξεις, γεγονότα έχετε να προσφέρετε ώστε να πείτε ότι δεν τρέχει τίποτα. Για δε την επιστολή, όποιος τη διαβάσει, νομίζω διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ψήγμα κάποιας αντίληψης ότι ήταν λάθος αυτή η συμπεριφορά κάποιας προσπάθειας για αποκατάσταση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παραβίαση ρητή του άρθρου 21.1 του SWIFT που οδηγεί στην ε, ε, πάυση της λειτουργίας του, στην ανέρεσή του. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μιλήσετε για καταγγελία που θα προτιμούσα εγώ τη ε, συμβάσεω ή μη τι άλλο, πρέπει να αναλογιστείτε το πάγωμα, την άρση αυτή τη συμφωνία. Το οφείλουμε αυτό στου Ευρωπαίου. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω σπουδάσει νομικά και είμαι βεβαία ότι όταν κάποιος παραβιάζει τον νόμο πρέπει να βλέπει και τις σχετικές συνέπειες. Όταν λοιπόν έχουμε παραβίαση ε, κανόνων στην Ευρώπη, προσβολή δικαιωμάτων των πολιτών ή των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αυτό δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο. <laughs> Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην έκθεση έκαινου την οποία είχαμε η οποία έχει συνταχθεί πριν από τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και όπου ήδη καταγγέλλονταν οι παρακολουθήσεις, οι παράνομες από πλευράς των υπηρεσιών των ΗΠΑ εις βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είδα να ευωδώνεται αυτή η έκθεση. Το Κοινοβούλιο εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον ασχολείται με τις ε, ε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στον Κουαντάναμο ενδιαφέρεται για τις σχέσεις και συμμαχίες με κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που συνέπραξαν στους βασανισμούς αυτών των κρατουμένων. Έχει βγει τίποτα από όλα αυτά. Όχι. και όταν κάποιος τόλμησε και έδωσε πληροφορίες δημόσια ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη σε όλο τον πλανήτη, είναι δυνατόν τα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα να μην έχουν καμία ένομη συνέπεια. Δεν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι παραβιάσεις αυτών των κανόνων να έχουν συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και Πάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Αλλά θα περάσω στο θέμα για να αναφερθώ στην αξία της συμφωνίας SWIFT που είναι και η καταπολέμηση τρομοκρατίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων ταυτόχρονα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως είναι δυνατόν πάνω σε αυτή τη συμβατική βάση να ε, γίνεται λόγος για διακοπή της λειτουργίας τους, δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα. Το Κοινοβούλιο είναι πεπισμένο ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε ε, η χρηματοδότηση, η οδή χρηματοδότηση ε, της τρομοκρατίας, σε αυτό δεν έχει αλλάξει τίποτα, το έχουμε δηλώσει απερίφραστα και δεν έχει αλλάξει τίποτα και γι' αυτό πιστεύω ότι η συμφωνία SWIFT θα πρέπει να ε, σταματήσει να λειτουργεί, να διακοπεί η λειτουργία της, να αρθεί, μόνο αν θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση να το πράξουμε μόνοι μα αυτό, την παρακολούθηση δηλαδή της χρηματοδότησης τη της ε, κατά τα άλλα, οποιαδήποτε προσπάθεια για πάγωμα, άρση λειτουργία και το καθεξής μας θέτει σε κίνδυνο. Και διερωτώ, γιατί κάποιοι ζητούν την άρση αυτή τη συμφωνίας πριν να έχουμε προχωρήσει, πριν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή, πριν να έχει ολοκληρώσει εργασίες σε αυτή η ομάδα που έχει θεσπιστεί. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα τη ομάδα εργασία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αποδεικτικά στοιχεία και η Επίτροπος δεν μας λέει ότι δεν έχει τηρηθεί η συνθήκη ή ότι το SWIFT δεν έχει προσφέρει ε, όσο όφιλε τον σεβασμό στην προστασία των δεδομένων. Δεν έχουμε δεδομένα δηλαδή και αποδείξεις, εκτός από αυτά που μας έχουν πει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σε αυτά πάλι, όσο έχω εγώ τουλάχιστον διαβάσει, γίνεται μια παραπομπή σε ένα χειρίδιο του, της NSA για την παρακολούθηση του SWIFT. Δεν έχουμε λοιπόν... Δύο φράσεις παρακαλώ. Ε, δεν έχουμε λοιπόν αποδείξει, αλλά έχουμε δύο διαφορετικές δυνατότητες δράσης. Είτε την νόμιμη, δηλαδή τη συμφωνία, την αξιοποίηση συμφωνίας, είτε την παράνομη. Λοιπόν, γιατί θέλουμε, γιατί θέλουν κάποιοι, όταν υπάρχει η νόμιμη συμφωνία ε, και η νόμιμη μέθοδος καταγραφής δεδομένων να την καταργήσουν για να καταφύγουμε τελικά στην παράνομη, στη μη νόμιμη παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων. Είτε έχει ε, ε, εφόσον δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι έχει κάνει κάτι το παράνομο η NSA και εφόσον δεν έχουμε ακόμα δικό μας σύστημα. Ένα λεπτό παραπάνω. Κύριε Βος, όμως η κυρία Ινφέλτ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση με την μπλε κάρτα. Yes, thank Κύριε όλοι εδώ αναφέρονται σε στοιχεία και αποδείξεις. Έχουν ε, προβληθεί πολλοί ισχυρισμοί για την ανάγκη και τη χρησιμότητα αυτών των στοιχείων ε, για την κατανόηση της τρομοκρατίας. Αυτοί οι ισχυρισμοί ε, δεν είναι βάσιμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ερώτησή μου είναι εξής. Η ομάδα σας και η κυβέρνησή σας θα υποστήριζε μια έρευνα από την υπηρεσία κυβέρνοχώρου του κυβερνού εγκλήματο τη ε, Europol. Γιατί κανένα μα δεν είναι εμπειρογνώμος και κανένα μα δεν έχει καταφέρει να δει μέσα στο SWIFT. Δεν θα έπρεπε να αφήσουμε το θέμα στα χέρια των εμπειρογνωμόνων τη πληροφορική για να πάνε επιτόπου και να κάνουν ε, μια έρευνα για το κατά πόσον έχει γίνει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία χωρί άδεια. Υποστηρίζετε αυτή την πρόταση. Yes, Mr. Voss. δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η κυβέρνηση από τη Γερμανία ή της Γερμανίας δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα περιστατικά. Γι' αυτό δεν είμαι σε θέση να αντιληφθώ το νόημα της ερώτησής σας και να δώσω απάντηση. Πάντως έχουμε κάνει ερώτηση στο SWIFT, έχουν στη θέση τους το know-how και έχουν απαντήσει ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τέτοια ίχνη τα οποία δεν εντοπίστηκαν όμως. Ε, η κυρία Νετφέλη δυστυχώς δεν ακούγεται δεν έχουμε στοιχεία και αν θέλουμε να, ε, να συμπεριφερθούμε κατά τρόπο αντίθετο με τους κανόνες αυτής της συμφωνίας, θα ήταν μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε την επιλογή είτε νόμιμη οδός είτε παράνομη. Αυτό είναι όλο. Η ε, κυρία Ζέπελ ανέφερε πολλές από τις ανησυχίε της ομάδας μου. Να ξεκινήσω με το θέμα της ε, διαρεύνησης ε, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βος. Εγώ ήδη έθεσα το θέμα της μονάδας της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του κυβερνού κλίματος και το Συμβούλιο ε, είπε ότι ε, μπορεί να κάνει μια τέτοια έρευνα και αν έτσι έχουν τα πράγματα, ένα από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το ζητήσει. Από εκεί πέρα, ε, το κατά πόσον θα γίνει η διαρρέμιση των διαρροών είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να διαρνήσουμε το τι συμβαίνει μέσω της συμφωνίας SWIFT. Ο κύριος Βος δεν με ακούει καν, εν πάση περιπτώσει. Ε, ελπίζω να μου δώσετε άλλο ένα λεπτό πρόεδρε μόλις γυρίσει ο κ. Βος. Εν πάση περιπτώσει. 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει γιατί στην έρευνα κανένας δεν ορ... καταθέτει με όρκο ε, οπότε ε, ξέρετε από εσάς κύριε Επίτροπε, να ε, πάρετε τις απαντήσεις και εσείς αναφέρετε, αναφέρεστε κατά βάση σε αυτή την έρευνα η οποία δεν μπορεί να δώσει σαφή αποτελέσματα. Ε, εμείς ε, δεν μπορούμε βέβαια να ακυρώσουμε τη συμφωνία, το Συμβούλιο μπορεί να την ακυρώσει με πλειοψηφία και η κυρία Ιντβέλτ έχει δίκιο. Ε, έχουμε ε, ε, εξουσία σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές συμφωνίες. Αυτό είναι ο μοχλός πίεσης που έχουμε και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οπότε να επαναλάβω ότι το SWIFT είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία για μας και για την ομάδα μας. Διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία αυτή στο Κοινοβούλιο, την πήραμε στα σοβαρά, καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις της και όλα αυτά τα παίρνουμε στα σοβαρά. Γι' αυτό το λόγο ε, θέλουμε η έρευνα να είναι όσο πιο λεπτομερής γίνεται, θα την αξιολογήσουν, θα αξιολογήσουν τα αποτέλεσματά της και τότε θα πάρουμε και μια πολιτική απόφαση για την αναστολή προσωρινή και ενδεχομένως αναδιαπραγμάτευση. Ε, δεν πρόκειται να είναι μια βιαστική απόφαση, η απόφαση θα είναι σοβαρή, αλλά θα είναι μια πολιτική απόφαση τελικά. Ευχαριστώ κύριε Μωράς. Ο συνάδελφος Μέγερ. Ευχαριστώ πρόεδρε το, η ελάχιστη χειρονομία που θα πρέπει να γίνει είναι η αναστολή της ε, συμφωνίας. Είναι η ελάχιστη χειρονομία, η ελάχιστη κίνηση. Είναι το ελάχιστο που απαιτούν από εμά οι Ευρωπαίοι για να προασπιστούμε ε, την ε, ε, κυριαρχία μας. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, πού πρέπει να φτάσουμε δεν καταλαβαίνω. Ε, είναι προφανές ότι αυτό πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατασκοπική δραστηριότητα που έχει γίνει ποτέ από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Όποιος δεν θέλει να το δει αυτό είναι δικό του πρόβλημα, αλλά πάντως είναι προφανή τα γεγονότα. Και μιλώ για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και τη Ατλαντικής Αμερικής. Ε, γιατί να ε, χρησιμοποιούμε ε, άλλα μέτρα και σταθμά για τις ΗΠΑ και αλλά για άλλες χώρες. Μην ξεχνάτε ότι η Βραζιλία ε, με τα ίδια στοιχεία που έχουμε εμείς, η Βραζιλία μόλις είδε την κατάσταση απέτησε από τον πρόεδρο Ομπάμα μία εξή και μία διόρθωση. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να απευθυνθεί στον υπεύθυνο. Ποιο είναι υπεύθυνο, ο πρόεδρο Ομπάμα. Και να του ζητήσει να λάβει τι ευθύνε του. Διότι αυτό πρόκειται για ένα ε, εγκληματικό, ε, πρόκειται για μια εγκληματική δράση σε εμά. Στη χώρα μου, αν κάποιο κατασκοπεύει, αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάμε όμω και πώ συνήθει αυτή η συμφωνία ότι πριν από μερικά χρόνια παράνομα οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τα δεδομένα SWIFT των τραπεζών των Ευρωπαίων πολιτών, τα αντλούσαν από εκεί και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να τιμωρήσει για αυτήν την ε, συμπεριφορά ε, επένεσε, ε, έδωσε και ανταπόδοση, δηλαδή νομοποίησε αυτή την, με τη συμφωνία αυτή τη συμπεριφορά. Ε, Προφανώ λοιπόν και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να πω ότι μάλλον θα πρέπει να καταγγελθεί αυτή η συμφωνία από αυτά που βλέπουμε. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει όμω η ειλικρίνεια σε αυτήν την υπόθεση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να ξέρουμε ότι με την άρση αυτή τη συμφωνία και με την Ερευνητική Επιτροπή που έχουμε στο Κοινοβούλιο, με την υποψηφιότητα του Σνόουντεν, για το βραβείο Ζαχάροφ. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι εν τέλει. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν υποβιβαστεί σε αντικείμενα προσωπικών δεδομένων, τα οποία αυθαίρετα μπορούν κάποιες αρχές να παρακολουθούν και να συλλέγουν. Χάνει την αξιοπρέπειά του ο άνθρωπος, χάνει το ε, καθεστώς του ως υποκείμενο δικαίου. Γίνεται ένα αντικείμενο και ζει μέσα στο φόβο και εν τέλει μέσα στην αυθαίρετη ε, απουσία εμπιστοσύνη. Τι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ένα όρομα, ένα όραμα μεγάλο όσο το, το φεγγάρι, ένα όραμα γεμάτο ε, μεγάλο όπως ο κόσμος ολόκληρος, όπως η ανακάλυψη της Αμερικής, ένα όραμα που δεν θα το εξαντλήσουμε σε μια ερευνητική επιτροπή, αλλά σε, στην απάντηση που θα δώσουμε στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι η διακυβέρνηση στο ίντερνετ, οι υποδομές, η προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων και η έρευνα η οποία θα κάνει σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα. Ε, αν δεν γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση δεν θα έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα <clears throat> και δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο για το γεγονός ότι ε, έχει τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης. Ε, έχει μιλήσει με τους Αμερικανούς και νομίζω ότι η κυρία Μάλστρομ παρακολουθεί από κοντά ε, το θέμα. Είμαι κάπως εξοικειωμένος με την ιστορία του TFTP. Ξέρω ότι οι Ολλανδοί πολίτες ανησυχούν πάρα πολύ για τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν. και οι συζητήσεις μας με τους εκπροσώπους του NSA δεν κάνουν πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Θα πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογή της συμφωνίας. ούτως ώστε να περιλαμβάνει ε, τα πάντα. Ε, αν περιοριζόμαστε μόνο στην καταπολέμηση ε, της τρομοκρατίας, ίσως περιορίζουμε κάπως το πεδίο εφαρμογής. Τι γίνεται με τα οικονομικά προβλήματα. Ε, νομίζω ότι μιλάμε για ανείχνευση, για παρακολούθηση ε, και για διάφορες άλλες ε, ε, λειτουργίες. Θα πρέπει να γίνονται βέβαια σεβαστά διάφορα δικαιώματα, ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την διεθνή τρομοκρατία, αλλά έχουμε και οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, τις οποίες και αυτές θα πρέπει να τηρούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ανεξάρτητα του τι έχει ψηφίσει ο καθένας για την ε, συμφωνία TFTP, ε, σε μια συζήτηση στην οποία αναφέρεται συνεχώς η ανάγκη να βασιστούμε στα στοιχεία υπάρχει κάτι που δημιουργεί σύγχυση γιατί το Κοινοβούλιο προσπαθεί να βεβαιώσει, να βεβαιωθεί για τα στοιχεία, εκπροσωπώντας εκατομμύρια πολίτες που ανησυχούν. Από την άλλη μεριά όμως μας αρνούνται το δικαίωμα να διαρμηνήσουμε τα γεγονότα. Παρόλε τις προσπάθειες της Κομισιόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Εθνική ε, Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν ε, ε, ε, δεν αρνήθηκε ότι έλαβε στοιχεία του SWIFT μέσω οδών που δεν είναι οι νόμιμες. Αυτό, αυτή η, παραδοχή και μόνο ε, ρίχνει σκιά στην, ε, στο κατά πόσον οι νομές Πολιτείες σέβονται τη Συμφωνία SWIFT. Η, Επιτροπή Έρευνας έδωσε την ευκαιρία στι ΗΠΑ να διαψεύσουν αυτή την ε, ε, περίπτωση, αυτό το σενάριο και δεν το έκαναν οι ΗΠΑ. Ακόμα και οι υπηρεσίες του SWIFT δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν σίγουρα ότι τα συστήματα ελέγχου τους δεν παραβιάστηκαν από μια κυβερνό επίθεση εκ μέρους της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε η ερώτηση είναι, η Κομισιόν έχει σκεφτεί την δυνατότητα εν ώψη μιας τέτοιας σαφούς παραβίασης συνθήκης να ε, ε, να προσφύγει ε, εναντίον των πολιτιών προκειμένου να σταλεί η συμφωνία SWIFT. μια λογική ανησυχία δημιουργείται από όλε τι ειδήσει που ακούμε περί ενδεχόμενης μαζικής παραβίασης των ε, θεμελιών δικαιωμάτων μέσα των ΗΠΑ. Η Κομισιόν νομίζω θα πρέπει να συλλέξει τι απαραίτητε πληροφορίε, έτσι ώστε ε, να προβάλλουμε μια ενιαία στάση ε, και αυστηρή στάση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, προσωρινά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Όμω αυτό το επεισόδιο κυρίω θα πρέπει να, χρησιμο... να χρησιμεύσει έτσι ώστε να ενισχυθεί η νομοθεσία προστασία των δεδομένων και ε, ο ιδιωτικό χαρακτήρα των ε, ε, συνομιλών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών αν ο, η, ο ε, ε, αν κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα επικράτησε η ιδέα ότι οι πόλεις μας καθιστούν ε, πιο ελεύθερους ε, πιο ελεύθερους από το φεουδαρχικό σύστημα της τους έτσι και σήμερα ο ευρωπαϊκός αέρας θα πρέπει να εγγυηθεί την, την ατομική μας ζωή ε, ο αέρας της ελευθερίας από, από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιτεθεί στους ανέμους που προσπαθούν να σηκώσουν διάφορες σκοτεινές δυνάμεις. Πρόεδρε, Εν ολίγη, η συζήτηση αυτή μα δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα τη πρόσβαση ε, στα δεδομένα προκειμένου να αποτρέψουν σοβαρά εγκλήματα εις βάρος ε, των ε, ε, Ευρωπαίων πολιτών, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν θέλει να χορηγήσει ε, λευκό επιταγή για την πλήρη παρακολούθηση των ε, συναλλαγών που προσπαθούν ως συνήθως οι μυστικές υπηρεσίες να εξασφαλίσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεμοφύλακας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών και εδώ έρχεται να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Αυτό λοιπόν ξεπερνάει την απλή αποστολή επιστολών, την καταγραφή διαμαρτυριών και καταγραφή ε, δεδομένων. Πρέπει η προστασία της προσωπικής ε, σφαίρας, του ιδιωτικού βίου δηλαδή, να εξασφαλιστεί κατά τρόπο ώστε να μην χορηγηθούν πλέον άλλα δεδομένα στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα SWIFT πρέπει να ε, ανασταλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει βέβαια να θυσιάσει όσο σημαντικές και αν με, την Ευρωπαϊκή, με τις ΗΠΑ, στο βωμό αυτών τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να πάψουμε να κάνουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Θα πρέπει να πάψουμε να συμπεριφερόμαστε όπως το παρελθόν. Και θα πρέπει να δείξουμε ότι διαφωνούμε με αυτή την συμπεριφορά των ΗΠΑ και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να είναι στο, για το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι τέτοιο. Πρέπει να δείξουμε τι εννοούμε, πρέπει να δείξουμε τι σημαίνει αυτό που θέλουμε για να το καταλάβουν και οι Αμερικανοί. Uh, Καλώς συνεχίζουμε με τη διαδικασία Καρστιάε και πρώτος το λόγο θα πάρει ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι για ένα τόσο λεπτό θέμα ίσως θα πρέπει όχι να χρησιμοποιούνται μεγάλα πολιτικά επιχειρήματα, ε, αλλά να περιοριστούμε στην κοινή λογική. Έχουμε να κάνουμε μια καταγγελία πιθανής κατασκοπίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε μία έρευνα για να επαληθεύσουμε αν υπάρχει πραγματικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα ή όχι. Επίσης, ισχύει η αρχή της προφύλαξης. Όταν υπάρχει ε, υποψία, αναστέλλεται η συμφωνία για την οποία ε, συζητάμε. Αν τελικά η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε πραγματικά για παραβίαση ε, λεπτών ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, τότε θα πρέπει να θέσουμε Λοιπόν, συζήτηση τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Εγώ δεν βλέπω καμία εναλλακτική λύση σε αυτή την απλή αλυσίδα ε, δράσεων. Έρευνα, αναστολή εντωμεταξύ και όταν επαληθευθεί ε, η υποψία, καταγγελία της συμφωνίας. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ο κόσμος έχει σοκαριστεί από τις ε, αποκαλύψεις του Σνόουντεν. Μάθαμε ότι η NSA ε, κάνει βιομηχανική κατασκοπία κατά της Βραζιλίας, ε, πολιτική κατασκοπία εναντίον πολιτικών ηγετών και των συναντήσεών τους, καθώς επίσης και παρακολουθεί κοινούς πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά δεν είναι αρκετά ώστε να συμφωνήσει η Επίτροπος να αναστείλει τη συμφωνία ως ότου ολοκληρωθεί μια ε, περιστατωμένη έρευνα. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Mr. Engstrom, colleague Pasca. Συνάδελφος Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με τους συναδέλφου Οι διαπραγματεύσεις, οι προτάσεις για τις δραστηριότητες της NSA πρέπει να είναι ψύχρεμες, όχι ιστερικές. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και δεδομένα και σε διαπιστώσεις σχετικέ με την ενδεχομένη παραβίαση δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστολή του Υπουργού Κόεν δεν μπορεί όμω να αντικαταστήσει τι ε, ενέργειε των ερευνητικών μας αρχών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τις αρχές της Europol να επαληθεύσουν τους ισχυρισμού και τα δεδομένα που ακούγονται και αναλόγως να ενημερώσουμε τους Αμερικανούς εταίρους κυρία Πρόεδρε, η αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτη. Ο πολίτης και κυρίως ο νεαρός πολίτης της Ευρώπης είναι όλο και πιο ενήμερος για το τι συμβαίνει. Ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις μας. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Κύριε Στογιάννευ, ε, δεδομένου του, της ύπαρξης, δεδομένης ύπαρξης ε, εξτρεμιστικών κινημάτων στον κόσμο πρέπει να δούμε τι γίνεται και από την άλλη μεριά ε, του Ατλαντικού ωκεανού. Υπάρχει ένα σύστημα γεστάπο που κατασκοπεύει συνεχώς τους πολίτες ε, δεν είναι επιλογή των Αμερικανών αλλά ε, επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όταν αυτά τα ζητήματα όμως χρησιμοποιούνται και εναντίον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Γινόμαστε ολοκληρωτικό καθεστώς με πολλή ασφάλεια και λίγες ελευθερίες. Γνωρίζουμε τέτοια καθεστώτα. Ε, εγώ έχω ανάγκη περισσότερη ελευθερία και όχι τόσο πολύ την ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταγγείλουμε τη SWIFT. Κυρία Επίτροπε. Um, η συμφωνία TFTP είναι μια διεθνή συμφωνία την οποία διαπραγματευτήκαμε. Ορισμένοι από εσά δεν υπερψηφίσατε, δεν σα άρεσε. Δικαίωμά σα. Ορισμένοι από εσά ψηφίσατε ναι, αλλά ε, χωρίς πολύ ενθουσιασμό. Αλλά η συμφωνία υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Διαπραγματευτήκαμε σημαντικές ε, σαφείς κανόνες για τη διαφάνεια, για το ποιος έχει πρόσβαση κλπ. Και επανεξετάσαμε τη συμφωνία και είδαμε ότι τη χάνει σεβασμού, υποβλήθηκαν προτάσεις για βελτίωσή της και έγινε και μια μελέτη αξιολόγησης για την χρησιμότητα του συστήματος. Αυτή η έκθεση είναι έτοιμη, δεν την έχω δημοσιοποιήσει, προκειμένου να γίνει πρώτα αυτές οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ε, σύντομα όμως θα την δημοσιοποιήσουμε. Και θα δείτε ότι η μελέτη δίνει σαφή ε, αντίρρητα, αντίρρητα στοιχεία ότι είναι χρήσιμη, χρήσιμο το σύστημα και για τις πολιτείες και για την Ευρώπη για την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Τώρα, ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτή η συμφωνία, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν μπορούμε να ε, αναστείλουμε μια συμφωνία με βάση ειδήσει, ειδησιογραφικές πληροφορίες. Οι ισχυρισμοί ήταν επαρκή έτσι ώστε να θέσουμε ερωτήματα στις Πολιτεία. Έστειλα επιστολέ, μίλησα τηλεφωνικά μαζί τους και συναντήθηκα με τον κύριο Κοέν ε, επί μακρόν τη Δευτέρα. Μου απάντησε πολλές ερωτήσεις, ε, πρέπει να τεθούν ακόμα και άλλες ερωτήσεις ε, και πιστεύω ότι η Επιτροπή Ελευθεριών θα θέσει αυτά τα ερωτήματα στην Ουάσιγκτον και ελπίζω θα πάρει και απαντήσεις. Ε, έχει γίνει σαφές ότι δεν έγινε παραβία συμφωνίας, δεν ε, έγινε κατευθείαν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του SWIFT στην Ευρώπη και ζήτησα αυτή η απάντηση να μου δοθεί και γραπτός. Ε, τώρα, συζητήσαμε και τα, τις, τους άλλους τρόπους πρόσβασης. Υπάρχουν άλλα format SWIFT που χρησιμοποιούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίω. Αυτό αναφέρεται και στο προήμιο της συμφωνίας μας και δεν καλύπτονται από τη συμφωνία SWIFT, για παράδειγμα. Το φόρμα SWIFT από τρίτη χώρα που γίνεται έρευνα και ενημερώνεται η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας ε, των ΗΠΑ ε, για συνήθεις αστυνομικές έρευνες. Αυτά, αυτές οι, ε, μεταβάσεις δεδομένων δεν καλύπτονται από SWIFT. Προσπαθώ να διευκρινίσω ότι δεν έρχονται σε αντίφαση με την TFTP αυτές οι, ε, πράξεις. Ο κ. Κοέν μου είπε επίσης ότι οι ε, αξιωματούχοι της NSA ε, εκπαιδεύονται για το πώς λειτουργούν τα τραπεζικά συστήματα και το πώς ερμηνεύονται τα μηνύματα SWIFT, αλλά με επιβεβαίωσε ότι δεν εκπαιδεύονται για παράνομη πρόσβαση στοιχεία του SWIFT. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Περιμένουμε ακόμα μερικές διευκρινήσει και γραπτός και ταυτόχρονα έχουμε και την πιο ευρία δουλειά που γίνεται σε διάφορε ομάδε εργασίας, στη δική σα στι επιτροπέ έρευνα, στην αντίστοιχη επιτροπή της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Συνεργαζόμαστε και με τη Λιθουανική Προεδρία στο πλαίσιο της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων. Και εγώ ανησυχώ για τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των Ευρωπαίων πολιτών. Γίνονται συζητήσει και ελπίζουμε ότι αυτό θα μα οδηγήσει σε συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορούμε να ε, βελτιώσουμε την προστασία των δεδομένων για του Ευρωπαίου πολίτες. Επίσης παρακολουθούμε πολύ στενά τα όσα λέει ο κ. Ομπάμα. Ε, ε, προσπαθεί και αυτό να ζητήσει υποστήριξη από το Κογκρέσο για να ρυθμίσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργία τη NSA. Αλλά πάντω μέχρι τώρα ε, οι επαφές μας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχουν ε, δώσει ενδείξεις για παραβίαση της συμφωνίας SWIFT. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνώ με την αναστολή της συμφωνίας. Ε, dear Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία κυρία Ενφιάς. Η συζήτηση αυτή έχει ολοκληρωθεί. Να σα υπενθυμίσω ότι το σχετικό ψήφισμα θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλη, τη δεύτερη του Οκτωβρίου.